Καλημέρα, συνάδελφοι. Ας ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία σήμερα το πρωί, όπως ε, φαίνεται στην ημερήσια διάταξη. Ε, αυτό γίνεται επισήμω υπό την ευθύνη τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Χθε ε, ε, η Επιτροπή επεξεργάστηκε το σχέδιο έκθεση και τι τροπολογίε. Ο κύριο Ευγέννη Κυρίλοφ, ο εισηγητή, θα θέλει να πει κάτι πριν ξεκινήσουμε. Κύριε Κυρίλοφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με τη συζήτηση χθε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η στρατιωτική ε, διάσταση του ε, ευρωπαϊκού έργου ενιαίας ενιαίου ουρανού ε, μας κάνει να έχουμε μια σωστή προσέγγιση στον τομέα αυτό και θα το υποστηρίξω γιατί δεν υπάρχουν αντιφάσεις όσον αφορά στις τροπολογίες ή σε δυσκολίες ε, με κάποιες συγκεκριμένες ιδέες. Έχουμε μια καλή υποστήριξη. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι η Επιτροπή ε, Μεταφορών να λάβει υπόψη της και να εγκρίνει όλες αυτές τις αλλαγές, γιατί λόγω της στρατιωτικής ε, διάστασης μπορεί να καθυστερήσει το project και να σέρουμε τα και να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ξεκινάμε λοιπόν τις, ε, την ψηφοφορία. Τροπολογία 1 του κυρίου Λίσεκ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία του κυρίου Λούχαν. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην παράγραφο 5, το πρωτότυπο, και έχουμε χωριστή ψηφοφορία σε τρία μέρη. Μέρος 1, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Μέρος 2, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Μέρος 3, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι επόμενες τρεις καταπίπτουν προφορική του δύο του κυρίου Λίζα κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 του εισηγητή υπέρ, 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην προφορική τροπολογία 3 του κυρίου Γκάλερ, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 του εισηγητή, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 4 του κυρίου Λούχαν, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Νούμερο 10, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και νούμερο 12 του κυρίου Γκάλερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ηλεκτρονικά ψηφίζουμε το σχέδιο της νομοδότησης όπως πετροποποιήθηκε. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται με πλειοψηφία 34, 34 ψήφων και δύο αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Κυρίλοφ. So we continue with the SEDE uh, draft agenda. Συνεχίζουμε με την ε, ημερήσια διάταξή μας. Bien, chers collègues. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Συνεχίζουμε τις εργασίες της υποεπιτροπής μας. Με τρία κείμενα. που αφορούν τις προτάσεις ε, Ορίζον 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που αφορά το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη για την περίοδο 2014 με 2020. Έξι προτάσεις περιλαμβάνει το πακέτο αυτό και η υποεπιτροπή μας όπως και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων αποφάσισαν να γνωμοδοτήσουν για τις τρεις πρώτες προτάσεις ε, που έχουν ε, αντίκτυπο στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή Ήτρε είναι αρμόδια επί της ουσία. Ο κύριος Μαυρονικόλας, ο κύριος αντιπρόεδρός μας, είναι ε, συντάκτης νομοδότησης και του δίνω το λόγο για να μας πει τα πρώτα του σχόλια για το πακέτο αυτό. you, President. I will discuss... Ευχαριστώ πολύ. Θα αναφερθώ και στις τρεις γνωμοδοτήσεις ε, και στις τρεις μαζί. Ε, η έρευνα και η ανάπτυξη είναι σημαντικό τμήμα του ορίζοντα 2020 και υπάρχει επίσης και η πρόκληση ε, συνεκτικής και ε, καινοτόμου οικονομίας ε, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις αυτές. Όσον αφορά τη νομική βάση και τις ηθικές βάσεις του ορίζοντα 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο επιβάλλει τις αξίες αυτές στην αξιολόγηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στην έρευνα για τα θέματα της ασφάλειας. Όλες αυτές οι δραστηριότητε υπό τον ορίζοντα 2020 δεν θα έπρεπε να επικεντρωθούν αποκλειστικά σε ε, πολιτικά σε τομεί πολιτικού, ε, γιατί υπάρχουν όλο και περισσότερε διτέ εφαρμογέ και όλο και περισσότερη συμπληρωματικότητα παρατηρείται μεταξύ τη ευρωπαϊκή άμυνα ε, και τη έρευνα των προβλημάτων ε, του στρατιωτικού τομέα. Αναφέρεται συγκεκριμένα στο άρθρο 6 ότι η έρευνα και η καινοτομία και οι σχετικές δραστηριότητες υπό τον ορίζοντα 2020 θα επικεντρωθούν κυρίως στις ε, πολιτικές εφαρμογές. Στον παράγραφο 2 ε, θα υπάρξει τροπολογία με διαφορετική διατύπωση ώστε οι στρατιωτικές εφαρμογές στο πλαίσιο της διτής χρήσης δεν θα αποκλείονται. Υπ' αυτήν την έννοια θα ήθελα να τονίσω τη σημασία τη δομή και τη εφαρμογή του ορίζοντα 2020. Σε σχέση με τις ε, προκλήσεις ε, της κοινωνίας ε, υπάρχουν τάσεις αντιμετώπισης των προκλήσεων που αντιμετωπίσουμε σήμερα, όμως υπάρχει αμφιβολία όσον αφορά το συντονισμό των δραστηριότητων στο πλαίσιο τη πρόκληση που υπάρχει πλέον για την γενοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη. Ίσως θα πρέπει να υπάρχει μια υποδιέρεση μεταξύ των συνεκτικών κοινωνιών και των ε, ε, καινοτόμων κοινωνιών και από την άλλη ε, των ασφαλών κοινωνιών. Αυτή η ιδέα προέρχεται από, τον εισηγητή, από την κυρία Μαντουρέλ, την εισηγήτρια στην Ήτρε και συμφωνούμε επ' αυτού γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στην πτυχή της ασφάλειας και της άμυνας η πρόληψη είναι επίσης πολύ σημαντική για να μπορούν οι κοινωνίες να προλαμβάνουν ε, ε, σε οποιαδήποτε κρίση και πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να προβαίνουν σε έρευνα ε, για την ασφάλεια ε, η οποία πρέπει να διατηρηθεί ως σημαντικό τμήμα του ορίζοντα 2020 και η εμβέλεια, το πεδίο εφαρμογής θα έπρεπε να επεκταθεί για να συμπεριλάβει την ανάγκη μεταφοράς τεχνογνωσίας και καινοτομίας... μεταξύ ε, του πολιτικού και του στρατιωτικού τομέα. Για τον ορίζοντα, ορίζον 2020 θα έπρεπε να υποστηρίζει ε, την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 42.2 και στο άρθρο 45 της ε, Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα αυτό θα έπρεπε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσει διτής χρήσης ε, της έρευνας και της καινοτομίας και οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να ε, δημιουργήσουν υποδομές για τη σταθερότητα, την ασφάλεια, την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, όπως επίσης και για τη διαχείριση των κρίσεων. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας πρέπει να αναγνωριστεί, γιατί μπορεί να είναι ένας από τους βασικούς σετερούς για, ε, περαιτέρω, για περαιτέρω συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας. Ο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, Άμυνας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του καθήκοντος που του έχει αναθέσει το Συμβούλιο μπορεί να κληθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις ε, για συνεργασία σε, συγκεκριμένες, ε, σε συγκεκριμένους τομείς όπως για παράδειγμα η εσωτερική αγορά, η έρευνα, η ανάπτυξη, η καινοτομία κλπ. Είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο της διάδοσης ε, στο πλαίσιο του ε, ορίζοντα 2020 για την προστασία της ελευθερίας και της σταθερότητας ασφάλειας ε, των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πρωτοστατήσει και να ενισχύσει ε, ε, τους ε, διάφορους τομείς προς την κατεύθυνση της καινοτομίας. Είναι πολύ σημαντική η προετοιμασία και η πρόληψη των ε, απειλών στην ασφάλεια. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προκλήσεις που δεν μπορεί να δοθεί σε ανεξάρτητους τομείς. Ε, χρειάζεται συντονισμένη, σφαιρική και φιλόδοξη προσέγγιση. Η έρευνα και η καινοτομία είναι μεγάλη σημασία ε, για την έρευνα και την ασφάλεια και δείχνει και τη σημασία ε, της ε, ασφάλειας για την ε, επίτευξη των στόχων του ορίζοντα 2020. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκόμες. Να πω απλώς ότι υποστηρίζω πλήρως αυτά που είπε ο κύριος Μαυρονικόλας. Είναι μια ε, ολοκληρωμένη προσέγγιση και πραγματικά είναι ένα κεντρικό θέμα. Όσοι εξημών ε, ζητούμε και καλούμε για περισσότερη Ευρώπη, κυρίως ε, στον χώρο της ασφάλειας και της άμυνας, δεν μπορούμε παρά να υποστηρίξουμε αυτά που είπε. Και αυτό μπορούμε να το μεταφράσουμε σε δράση μέσα από αυτές ε, τις εκθέσεις για τον ορίζοντα 2020, γιατί αυτό είναι το μέλλον. Έχει να κάνει να βάλουμε τα χρήματά μας εκεί που πρέπει, υποστηρίζοντας με χρηματοδότηση όχι μόνο τις δραστηριότητες έρευνας, αλλά και συγκεκριμένες εφαρμογές, αυτές εφαρμογές οι οποίες είναι διτής χρήσης οι περισσότερες και δεν πρέπει να αποφασίζουμε ποια είναι η στιγμή ξεκάθαρα να ε, πατάξουμε την αντίσταση κάποιων κρατών μελών τα οποία τώρα σε περίοδο κρίσης βλέπουν τα πλέον εκτήματα, αλλά δεν δίνουν τα χρήματα ούτε για την έρευνα, ούτε για τις εφαρμογές. Και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά από τα πράγματα που στη θεωρία υποτίθεται ότι είναι η δουλειά μας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω και στο γεγονός ότι έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε στη διάδοση αυτών με, στους ενδιαφερόμενους, ε, γιατί υπάρχει μια βιομηχανική βάση στην ασφάλεια και στην άμυνα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εμπλεκόμενοι κατανοούν τις δυνατότητες που προσφέρονται από την συμπερίληψή τους σε αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο ορίζοντας 2020. Και οι ίδιοι προφανώς θα σκίσουν και πιέσεις στις κυβερνήσεις μας για να το αποδεχτούν. Νομίζω ότι ο ρόλος του φορέα αυτού, όπως είπε ο κύριος Μαυρονικόλας, είναι πολύ σημαντικός. Στην Πορτογαλία, με την κυρία Μαρία Γκράσα Καρβάλο, που είναι η συγκήτρια για την Ήτρε, κάναμε μια δημόσια ακρόαση με τους εκπροσώπους του φορέα αυτού, του ΕΟΑ συγκεκριμένα για να μπορέσουμε να επιστήσουμε την προσοχή των ενδιαφερομένων και των οργάνων της κυβέρνησης ε, για αυτό το θέμα. Νομίζω λοιπόν ότι στην Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις προτάσεις του κυρίου Μαυρονικόλα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κρούνμπαρκ. Thank you, Chairman. I would be opposed to including the military. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ αντιτίθαμε στην συμπερίληψη της ε, στρατιωτικής χρήσης και υποστηρίζω την αποκλειστική χρήση για πολιτικούς σκοπούς για τον εξή λόγο. Μιλάμε για μεταφορά τεχνολογίας και ανταγωνιστικότητας. Στο παρελθόν υπήρχε ιδέα ότι η, ως προς την δυτή ε, χρήση ε, θα είχαμε πρώτα την στρατιωτική ε, διάσταση και μετά θα διαδίδαμε την τεχνολογία στην ε, ε, μη στρατιωτική διάσταση. Σήμερα γίνεται το αντίθετο. Από την άλλη, το να έχουμε και τις δύο μαζί και να ξεκινάμε με τις μη στρατιωτικές ε, χρήσεις της τεχνολογίας, αυτό υποστηρίζει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα με έναν τρόπο πιο αποτελεσματικό από το να προσπαθούμε να μοιραστούμε τους πόρους εξ αρχής μεταξύ της στρατιωτικής και μη στρατιωτικής διάστασης. Άρα ε, σήμερα ε, πάμε από τη μη στρατιωτική στη στρατιωτική διάσταση, γι' αυτό υποστηρίζω μόνο την πρώτη. Ε, δεν μιλάμε τώρα μόνο για pooling, αλλά για pooling και sharing. Έχουμε λίγες, λίγους στρατιωτικούς πόρους ε, και με τόσους λίγους πόρους είναι καλό να συγκεντρώνουμε, να κάνουμε pooling ε, και των ε, πόρων για την έρευνα. Αυτό θα λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά αν δεν δώσουμε χρήματα για, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να αφήσουμε αυτό το, αυτή τη συγκέντρωση και το μοίρασμα να λειτουργήσει από κάτω προς τα πάνω. Υπάρχει επίσης ε, και μια ολόκληρη συζήτηση για το πώς χρησιμοποιούμε αυτούς τους πόρους. Έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση για την χρήση ε, αυτών των λίγων ε, πόρων που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης για το στρατιωτικό τομέα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι ε, αντίθετος με την ε, προηγούμενη ομιλήτρια, εγώ ε, θεωρώ ότι έχουμε ήδη συζητήσει αυτό το θέμα στην Επιτροπή μας εδώ πριν γίνει αυτή η νομοθετική πράξη, δηλαδή έρευνα, καινοτομία προς υποστήριξη των αποστολών της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Έτσι λοιπόν, ε, έχουμε εδώ project που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια αυτής της κοινή πολιτικής και θα πρέπει να υποστηριχτούν. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Επίσης θα ήθελα να σας αναφέρω αυτό που ήδη έχουμε ε, αποφασίσει στην έκθεση κρατήρια ε, άρθρο 42 ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία μεταξύ του οργανισμού και της Κομισιόν με σκοπό να ενισχυθεί η δυνατότητα διτών χρήσεων ώστε να έχουμε την πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για έρευνα που σχετίζεται με την ασφάλεια και για να έχουμε καλύτερη διαχείριση των συνεργειών μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών πόρων, ειδικότερα μέσα στα πλαίσια του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Επίσης, ε, καλοχωρίζει καλωσορίζει ε, τους σκοπούς του προγράμματος που έχουν να κάνουν με την εσωτερική ασφάλεια και αναγνωρίζει και την πραγματικότητα της ε, διαχείρισης κρίσεων και προωθεί την ε, ασφάλεια και, την έρευνα για την ασφάλεια και την άμυνα. Άρα υποστηρίζω να είμαστε συνεπείς ως προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζω ότι αυτό θα λάβει, θα αντικατοπτριστεί στην έκθεση και στην απόφαση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Ζέμκε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε κάποια στοιχεία που μου φαίνονται σημαντικά. Καταρχάς, η πρόταση που προετοιμάστηκε από τον συνάδελφο μου φαίνεται πολύ καλή, πολύ θετική. Βλέπουμε ότι το κείμενο αυτό γράφτηκε από κάποιον που γνωρίζει τον τομέα αυτό, που έχει μια πρακτική εμπειρία και που ήταν επικεφαλής της άμυνας στη χώρα του. Αλλά θα πρότεινα στο κείμενο αυτό να υπάρξει μια παράγραφος για την έκθεση του κυρίου Λίσεκ γιατί η έκθεση του κυρίου Λίσεκ μας έδειξε ότι η κρίση που δυστυχώς η Ευρώπη ακόμα γνωρίζει, αυτή η χρηματοπιστωτική κρίση, αρχίζει να αγγίζει όλο και περισσότερο τα κράτη και τη δυνατότητά τους ε, και όλες οι δυνατότητές τους αμφισβητούνται τώρα. Δεν θα να σας δώσω τώρα νούμερα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα τρία-τέσσερα τελευταία χρόνια οι αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη μειώθηκαν τουλάχιστον κατά 15%. Υπάρχουν μάλιστα κράτη όπου αυτή η μείωση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι, αν η οικονομική κατάσταση δεν αποκατασταθεί γρήγορα στην Ευρώπη, τα κράτη θα προσπαθούν συνέχεια να κάνουν περικοπές και θα βρεθούμε σε μια παράλογη κατάσταση. Δηλαδή, ενώ θα υπάρχουν όλο και λιγότερα κονδύλια στη διάθεσή μας, παράλληλα θα έχουμε παράλληλα πολλά προγράμματα έρευνας. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουμε πάνω από 10 προγράμματα έρευνας, στρατιωτική έρευνας, που τρέχουν παράλληλα. Σας ενθαρρύνω λοιπόν να σκεφτείτε αυτό το πρόβλημα. Αν έχουμε λιγότερα χρήματα, θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα και να τα επενδύσουμε στο μέλλον. Δεν θα πρέπει να, τα, να στοχεύουμε στην κατανάλωση μόνο. Θα πρέπει να υπάρχουν κονδύλια για την έρευνα. Ξέρετε σε τι φάση είμαστε σε σχέση με τη Ρωσία, την, την Αμερική και την Κίνα και τι δαπάνε που κάνουν για την άμυνα. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα σκεφτεί και να τα απεικονίζει αυτό το έγγραφο στο, στο διατακτικό του. Ευχαριστώ κύριο Λουράν. Η συμπερίληψη της ε, έρευνας για την ασφάλεια σε μια κοινωνία καινοτομία και ασφάλειας είναι μια πολύ καλή πρόταση. Από τη δική μου πλευρά η... θεωρώ ότι οι πολίτε δεν είναι μόνο στόχος ε, επίθεσης, αλλά ταυτόχρονα είναι και αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια. Έτσι λοιπόν, αυτός ο ορίζοντας 2020, ε, αυτό το πρόγραμμα, εκφράζει πολύ σαφώς την ανάγκη ανάπτυξη στον τομέα αυτό. Πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της ασφάλειας και μέσω της έρευνας και της καινοτομίας. Από την έκθεση αυτή μπορεί να προκύπτει η ανάγκη ε, να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και την εγκληματικότητα, να ενισχύσουμε την ασφάλεια των συνόρων, το θέμα της κύβερνο-ασφάλειας η αντοχή της Ευρώπης σε περίπτωση κρίσεων ή καταστροφών και βεβαίως έχουμε μεγάλη εμπειρία στους τομείς αυτούς. Και θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο που για μένα είναι σημαντικό. Το να βρούμε τους λόγους της ριζοσπαστικοποίησης των ανθρώπων ε, συνδέεται και με, την, ε, το σχεδιασμό κατάλληλων κοινωνικών πολιτικών για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την πρόληψη πριν την παρέμβαση. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να αναγνωρίσουμε τα pattern, τις συμπεριφορές. Θέλω να σας μιλήσω για τον εξελικτικό χαρακτήρα της σχέσης ε, ασφάλειας και τεχνολογίας και αμυντικής τεχνολογίας απ' την άλλη. Πρέπει να υπάρχει έρευνα και να αναπτύξουμε τεχνολογίες που έχουν δυναμικό εφαρμογής και στους δύο τομείς, και στο στρατιωτικό και στο μη στρατιωτικό. Θα πρέπει να ενισχύσουμε και τις μη στρατιωτικές και τις στρατιωτικές παράλληλες εφαρμογές και στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και στον τομέα του ελέγχου των συνόρων. Θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Δεν, <coughs> νομίζω ότι μπορούμε να προλάβουμε 100% τις απειλές, όλες τις απειλές στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, όποιες και αν είναι αυτές. Είτε φυσικής προέλευσης, είτε ανθρώπινης προέλευσης. Επομένως πρέπει να επικεντρώσουμε στην ενίσχυση της ικανότητας ανάκαμψης της Ευρώπης. Ανάκαμψης από τις κρίσεις, όποιες και αν είναι αυτές. Νομίζω λοιπόν ότι η δυνατότητα συμμετοχής τρίτων χωρών είναι μια άλλη πτυχή, πολύ ενδιαφέρουσα. Θέλω να την... Είναι καλό καταρχήν θέμα, αλλά στην έκθεση και στην πρόταση της Κομισιόν δεν αναφέρεται πουθενά ξεκάθαρα ποια είναι τα κριτήρια για τη συμμετοχή αυτών των χωρών, των τρίτων χωρών. Και μιλάω για το άρθρο 7 του κανονισμού. Το άρθρο 7 του κανονισμού λοιπόν, όπου λέμε μόνο ότι οποιαδήποτε νομική οντότητα ανάλο, ανεξάρτητα από την έδρα της μπορεί να συμμετάσχει. Αλλά δεν έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια συμμετοχής τρίτων χωρών κτλ. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τη συμμετοχή αυτών των νομικών οντοτήτων, για να το πω έτσι. που με την δουλειά που κάνουν, με τους στόχους που έχουν ή λόγω της έδρας τους μπορεί εν δυνάμει να απειλήσουν, την, ε, να παρεμποδίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της υπό το διεθνές δίκαιο. Αυτά είναι τα θέματα που ήθελα να αναφέρω και χαίρομαι πολύ που λαμβάνω μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Πιστεύω και ελπίζω η έκθεση αυτή να συνεισφέρει σημαντικά και να βελτιώσει τον τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Κράμπεργκ. Μία ερώτηση σύντομη προς τον κύριο Γκάλερ. Οι πόροι που θα χρησιμοποιηθούν Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα υποστηρίξουν την ΚΠΑ και δεν θα μπουν σε εθνικές τσέπες και θα εξαφανιστούν. Ε, δεν μπορεί να πάει στους εθνικούς ε, προϋπολογισμούς γιατί οι αποστολές της ΚΠΑ ε, δεν μπαίνουν καν ε, το μεγαλύτερο κομμάτι στον προπολογισμό των κρατών μελών. Ε, μόνο το προσωπικό ε, είναι αυτό που χρησιμοποιείται από τα κράτη-μέλη και μόνο τα διοικητικά έξοδα αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Ό,τι έχει να κάνει με το υλικό και με το σχεδιασμό αυτά είναι πράγματα που αναλύουμε με τις αποφάσεις μας. Κοιτάμε δηλαδή να δούμε τι χρειαζόμαστε για την εκτέλεση αυτών των αποστολών. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι μια προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν μπορεί να εξαφανιστεί στους εθνικούς ε, προϋπολογισμούς γιατί από τη στιγμή που ε, βρίσκουμε ε, υλικό για τις αποστολές, ε, αυτό πληρώνεται και από τους εθνικούς προϋπολογισμούς και έχει να κάνει με την έρευνα και την ανάπτυξη σε προηγούμενο στάδιο. Πρέπει λοιπόν ε, εμείς να παρακολουθούμε τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο τότε, σε εκείνο το προηγούμενο στάδιο και μετά όταν γίνεται η χρήση τότε μπορεί να γίνει σε εθνικό επίπεδο αλλά ε, δεν μπορεί να χαθεί πια. Αυτό το, έτσι το βλέπω εγώ. Ωραία. Σας ευχαριστώ για αυτές τις ε, παρεμβάσεις. Ο κύριος Μαυρονικόλας θέλει να κατάληξε κάποια συμπεράσματα. Πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων στο θέμα αυτό. Θα λάβω υπόψη τις ε, παρεμβάσεις όλων των συναδέλφων. Μην ξεχνάτε όμως ότι πρέπει να πείσουμε και την εισηγήτρια την κυρία Ριέρα Μαντουρέλ ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η παράγραφος με τα βασικά στοιχεία που προτείνουμε. Πάντως ε, αυτές οι προτάσεις πιστεύω θα δεχτούν από όλη την Επιτροπή. Η Κομισιόν θέλει να παρέμβει στο σημείο αυτό. Ναι, Πρόεδρε πολύ σύντομα να διευκρινίσω το χαρακτήρα της πρότασης της Κομισιόν. Γιατί νομίζω ότι οι ευρωβουλευτές... Εντάξει, ε, λογικό είναι να μην γνωρίζουν ακριβώς ε, τις διάφορες διατάξεις που υπάρχουν στα διάφορα σημεία του προγράμματος. Θέλω πολύ γρήγορα να υπενθυμίσω σε όλους ότι στο σημερινό πρόγραμμα πλαίσιο 7 έχουμε ήδη την ίδια πρόταση που αναφέρεται στην αποκλειστική μη στρατιωτική εστίαση σε ό,τι αφορά το τμήμα της έρευνας του προγράμματος πλαίσιο 7. Και αυτό δεν εμπόδισε την Κομισιόν να υιοθετήσει ετήσια προγράμματα εργασίας, όπου η, διτή χρήση, η τεχνολογία διτής χρήσης αναπτύσσεται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργασίας. Υπάρχει αυτό, έχουμε δει πολλές συνεργασίες σε τομείς όπως το CBRN, ε, ραδιοεπικοινωνίες, ανεπάνδρωτα συστήματα, ε, εναέρια και ε, τεχνολογίες επιτήρησης. Στο πρόγραμμα πλαίσιο 8 θα συνεχίσουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή αυτός ο όρος αποκλειστική α, μη στρατιωτική χρήση δεν είναι συμβατός με, το, με τη δυτή χρήση. Σημαίνει τεχνολογίες μη στρατιωτικές που ενδεχομένως έχουν εφαρμογή στο στρατιωτικό τομέα. Φυσικά δεν θα θέλαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε καθαρά αμυντικές τεχνολογίες. Πιστεύουμε ότι η καθαρά αμυντική έρευνα θα πρέπει να διεξάγεται αποκλειστικά μέσα στον τομέα και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας με προπολογισμού που έρχονται από τα κράτη-μέλη και δίδονται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα. Λοιπόν, προσπαθούμε να λαμβάνουμε γενικά υπόψη όλες τις εκθέσεις του Κοινοβουλίου και τη Λίζα και τα λοιπά και νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν απέχει πολύ μακριά από αυτό που προτείνει ο Ευρωβουλευτής σας, ο κύριος Μαυρονικόλας. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάλερ. Γι' αυτό ακριβώς εγώ και η ομάδα μου θέλουμε να διαγράψουμε ακριβώς αυτή τη φράση, με αυτή που λέει η αποκλειστική χρήση. Έτσι για λόγου για να είμαστε σίγουροι. Από την άλλη, δεν μιλάμε για αμυντική έρευνα, μιλάμε για κάτι που συνδέεται με την αποστολή μας ε, στα πλαίσια της ΚΠΑ. Γιατί ούτω ή άλλω και αυτό το, υπο... το συμφώνησαν οι υπουργοί και τα κράτη-μέλη, ότι θα έχουμε αποστολέ ΚΠΑ. Δεν μιλάμε έτσι γενικά για άμυνα, μιλάμε για αποστολέ που έχουμε συμφωνήσει στα πλαίσια τη ΚΠΑ. Και για να τι υποστηρίξουμε και να προωθήσουμε ακριβώς αυτή τη συμφωνία των Υπουργών θα πρέπει α, να χρησιμοποιήσουμε τον ορίζοντα 2020 ε, με τον σωστό τρόπο. Γι' αυτό πρέπει να διαγραφεί αυτή η φράση που σα ε, εντοπίζω και που σα ανέφερα προηγουμένω. Πολύ ωραία. Προτείνω λοιπόν να παραμένουμε εδώ στι 11 Ιουλίου στην επόμενη συνοδό μα, στην επόμενη συνεδρίασή μα θα κάνουμε μια συζήτηση για το σχέδιο του κυρίου Μαυρονικόλα και η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι η 12η Ιουλίου. Ωραία. Πάμε τώρα στο δεύτερο σημείο που είναι η έκθεση που την, περιμένουμε, που την περιμένουμε με ανυπομονησία του κυρίου Τάραντα για το ρόλο της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας σε περιπτώσεις κρίσεων που οφείλονται στο κλίμα, των, στο κλίμα και στις φυσικές καταστροφές. Είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει τα μάλα, όπου πραγματικά ζητούσαμε, είχε ζητηθεί να υπάρχει μια έκθεση της Επιτροπής μας. Ε, θα δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Τάραντ για να μας παρουσιάσει το κείμενό του. Thank President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε ένα σχέδιο κειμένου της έκθεσης. Θα προσπαθήσω να σας το περιγράψω. Να περιγράψω το πνεύμα και τις προτάσεις που εμπεριέχει. Και περιμένω βεβαίως τη συζήτηση που θα ακολουθήσει μετά την παρουσίασή μου και τα σχόλιά σας. Οι προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για να θέσουν το θέμα στον ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Ιούλιο του 2011 και στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων για το έγκλημα και τη διπλωματία ε, οδήγησε στο ότι ε, το κλίμα, οι σχέση με την άμυνα ε, μπαίνουν πιο κοντά στο... εστιάζουμε σε αυτό μάλλον, καθώς και σε απειλές τις μελλοντικές. Μέσα στα πέντε χρόνια που ακολουθούν, ε, στον τομέα του κλίματος, των φυσικών καταστροφών και τη σχέση με την άμυνα, έχουμε κάνει πολλά. Ε, ο λόγος αυτής της έκθεσης είναι να την ευθυγραμμίσουμε, να ευθυγραμμίσουμε μάλλον αυτό το σημείο και να γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις και δράσεις και να υπάρξει μια πολιτική συζήτηση. Και να προσπαθήσουμε να συγκεράσουμε να πείσουμε μάλλον διάφορους φορείς που δεν θέλουν να συνομιλήσουν ε, αυτή τη στιγμή για όλα αυτά τα θέματα. Παρά την χρηματοπιστωτική κρίση, πιστεύω ότι είναι κατάλληλη στιγμή για να το κάνουμε. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η κυρία Άστον ε, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να, να κάνουν αυτό που υποσχέθηκε η υπατή Εκπρόσωπος στην αρχή της θητείας της. Ένα κοινό έγγραφο της ε, Υπάρχει ένα κοινό έγγραφο από τον Ιούλιο του 2011 της Κομισιόν και τη Υπηρεσία Εξωτερική Τράση με τρει τάσει. Και το ένα λέγεται κλιματική αλλαγή και διεθνής ασφάλεια. Αυτό υπάρχει. Αλλά τώρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι να είμαστε πιο δημιουργικοί, να έχουμε περισσότερη πολιτική βούληση και να είμαστε πιο, πολύ πιο ενεργητικοί. Υπάρχουν προτάσεις και συστάσεις σε αυτή την έκθεση που έλαβα υπόψη μου στη δική μου έκθεση, αλλά γενικά προτείνω να πάμε ακόμα πιο μακριά. Οι προτάσεις λοιπόν στον πρώτο τίτλο ε, πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση και δράση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα κατάλογο με προκλήσεις και θα πρέπει να έχει ένα κατάλογο με όλες τις χώρες που είναι ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές, τη, όπως η Αρκτική, ο Αραβικός κόσμο, τα Ιμαλάια, το πλατό, ε, η Οροπέδιο του Θιβέτ κτλ. Ε, μιλάμε για ευάλωτε κλιματικές αλλαγές. Έτσι. Επίσης θέλουμε να έχουμε ένα κείμενο πολιτικής με τις βασικές αρχές, ε, κατευθυντήρες γραμμέ και μέσα που έχει η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας, ε, όπου θα εντάξουμε την διάσταση του κλίματος, όπως ακριβώς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διάσταση του φύλου. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει στο Συμβούλιο μια ομάδα εργασία ή στην Υπηρεσία Εξωτερική δράση που θα εξετάζει όλο το φάσμα ε, διαπλεκόμενων θεμάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και με την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια και τα μελήματα περιάμινας. Με συντονισμό με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ανάπτυξης δυναμικού τονίζουμε την ανάγκη να βρούμε συνέργειες και συνεργασίες, δηλαδή να έχουμε προγράμματα όπου θα, θα φέρνουμε μαζί όλα τα μέσα μας και θα τα χρησιμοποιούμε από κοινού, ανάλογα με τις ανάγκες. Επίσης, Θέλουμε να υπάρξουν προτάσεις για την εφαρμογή ενός αρχικού α, ταμείου, άρθρο 41.3 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ούτως ώστε να έχουμε τέτοια προγράμματα ε, συγκέντρωσης και από κοινού ε, του, δυναμικού που υπάρχει. Επίσης, το δεύτερο τίτλο, η ανάγκη για ένα νέο πνεύμα, στρατηγική και ενοιολογικές προκλήσεις. Θέλουμε να υπάρξει πίεση ούτω ώστε οι αρνητικές συνέπειες της ε, κλιματικής αλλαγής στην ε, ασφάλεια και στην άμυνα να ενσωματωθούν. Σε όλες τις ε, στρατηγικές των εγγράφων της ΚΕΠΑ και της ΚΠΑ και που θα αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό των επιμέρους πολιτικών και των αποστολών. Ζητά από την ύπατη εκπρόσωπο να εξασφαλίσει ότι η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και οι διάφορε μονάδε που ασχολούνται με πολιτικέ άμυνα και ασφάλεια λαμβάνουν σε υπόψη τι ε, πιο πρόσφατε εξελίξει του διακυβερνητικού πάνελ για την κλιματική αλλαγή, IPCC, ε, και άλλων επίση ε, πιο πρόσφατων αξιολογήσεων και εκθέσεων. Επίση, οι εμπειρογνώμονε για τα κλιματικά θα πρέπει να υπάρχουν σε όλου του φορεί τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση που θα ασχολούνται με την ανάλυση και την έγκυρη προειδοποίηση, όπω παραδείγματο χάρη το Κέντρο Situation Center. Επίσης ζητάει από, τα, ε, από τους φορείς ε, εξωτερικής υπηρεσίας, εξωτερικής δράσης να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών με την Κομισιόν ε, καθώς και με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει διαφανής πρόσβαση ε, σε όλες τις ε, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και σε ανθρωπιστικές οργανώσεις από τις δομές αυτές ε, που είναι στρατιωτικές και μη στρατιωτικές. Επίσης, ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επίσης Εξωτερική Δράση και την Κομισιό να εντάξει την, το θέμα της κλιματικής αλλαγής στην ΚΠΑ, ούτως ώστε να υπάρχει σταθερότητα στον ενεργειακό ανεφοδιασμό. Επίσης, προτάσεις στον τέταρτο τίτλο. Η ανάγκη για θεσμική δημιουργικότητα, μέσα και δυνατότητες. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη στα, στρατιωτικά τους δόγματα να εντάξουν το θέμα της κλιματικής αλλαγής και ειδικά όταν μιλάμε για φορείς που έχουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται και να καταπολεμούν φυσικές καταστροφές όπως παραδείγματος χάρη κινητά, νοσοκομεία, επικοινωνία και τεχνολογία επικοινωνίας, δομές επικοινωνίας κτλ. Ε, καλεί το Συμβούλιο και την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα να διερευνήσουν τι δυνατότητε δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού Σώματο Μηχανικών ε, που θα το επανδρώσουν και θα το εφοδιάσουν με όλες τι απαραίτητες δομέ μέσα στα πλαίσια αυτού του pooling and sharing, τη συγκέντρωση δηλαδή από κοινού, και, χρήσης του δυναμικού. Ζητάει επίσης να χρησιμοποιηθούν α, όλες οι δυνατότητες στα πλαίσια του επόμενου πολιετούς α, πλαισίου 2014-2020, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν όλες τις δυνατότητες που έχουμε για την εξωτερική παροχή βοήθειας. Επίσης, ε, οι αποστολές μας στις πιο προβληματικές περιοχές και χώρες να χρησιμοποιούνται ε, για να έχουμε και κάθε πληροφορία για τις επόμενα, τα επόμενα, για τις καταστροφές ή και οποιαδήποτε προβλήματα υπάρχουν. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική θέση που θα δημιουργηθεί από την ύπατη εκπρόσωπο ενός ειδικού για κλιματικές αλλαγές. Αυτές είναι οι βασικές ιδέες της έκθεσης. Προσπάθησα να είμαι διαφορετικός από τον τρόπο που τα γράφω στο κείμενο, γιατί είναι, μιλάμε για μια πολύ απαιτητική τώρα έκθεση. Κυρία Νέιτσκι, που είναι η σκιώδης εισηγήτρια του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ταράν για την ε, έκθεσή του σε σχέση με τον ε, ρόλο της κοινή ε, πολιτικής και άμυνας ε, στις φυσικές καταστροφές και στο κλίμα. Είναι ενδιαφέροντα αυτά τα πράγματα που είπε. Υπάρχουν σημεία επί των οποίων θα ήθελα να σχολιάσω. Θα υπάρξουν τροπολογίες σχετικά. Ο βασικός μου στόχος ως κοιόδης εισηγήτριας για το ΕΛΚ θα είναι να προσεγγίσω το κείμενο με πρακτικό τρόπο προσπαθώντας να ενισχύσουμε ήδη υπάρχοντα μέσα και πολιτικές αντί να δημιουργούμε νέα. Πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην ενίσχυση των δεξιοτήτων ε, και των ικανοτήτων του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάλυση του αντίκτυπου των ε, καταστροφών ε, στην εθνική και διεθνή ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σκεφτεί την ανταπόκριση στις διεθνείς προκλήσεις ασφάλειας που προκύπτουν από τις φυσικές καταστροφές που μπορούν να έχουν έναν αντίκτυπο στις εσωτερικές πολιτικές μας και στις εσωτερικές μας δομές. Και το σημαντικότερο, πιστεύω, ότι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα έπρεπε να υποκατασταθεί, αλλά να συμπληρωθεί από την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Θα ήθελα επίσης να να επαναλάβω την έκκλησή μου στα μέλη της Επιτροπής ε, να μην δουν τα πράγματα μόνο από το πλείσμα των πολιτικών ιδεολογιών, αλλά υπό έναν ε, πιο ρεαλιστικό τρόπο, με ένα πιο ρεαλιστικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο, ο κ. Μαυρονικόλα, εκ μέρου ε, των Σοσιαλιστών, αντικαθιστά τον κύριο Παλέτσκη. Εγώ εκπροσωπώ τον Γιούστας Παλέτσκης, ο οποίος επικροτεί την ε, προσπάθεια του ε, εισηγητή να βάλει στο επίκεντρο ε, της διαδικασίας τις φυσικές καταστροφές και την ενίσχυση της δυνατότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση κρίσεων και της ανοικοδόμησης σε περίπτωση κλιματικής ή φυσικής καταστροφής. Έτσι, η κοινή γνώμη ε, γνωρίζει και πάλι το θέμα του κλίματος ε, που είναι ένα ε, πολύ σημαντικό θέμα και έχει δημιουργήσει χρόνια μια οικονομική και φυσική απειλή. Το θέμα είναι πώς θα βελτιώσουμε την ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα μέσα που ήδη διαθέτει σε φυσικές καταστροφές. Πρέπει να μπορεί να υπάρχει και στρατιωτική και μη στρατιωτική ανταπόκριση υπάρχει και ε, καλή συνεργασία μεταξύ τους. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να δούμε πού υπάρχουν δυνατότητες και πού υπάρχουν κενά και να δούμε ποια μπορεί να είναι η προστιθέμενη αξία της στρατιωτικής χρήσης. Θέλουμε λοιπόν να συστήσουμε στα κράτη-μέλη να βελτιώσουν καλύτερα την, ε, ε, την άμεση ανταπόκριση και την άμεση ανάπτυξη των ευρωπαϊκών δυνάμεων γιατί σε μερικές περιπτώσεις ε, μπορεί να είναι και τμήμα μιας στρατιωτικής επιχείρησης κάτι τέτοιο και υποστρατιωτική διοίκηση. Η έγκυρη αξιολόγηση ε, και η ανάπτυξη των δυνάμεων αυτών σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ανταποκριθεί χρησιμοποιώντας τα καλύτερα μέσα ώστε να αναπτύσσονται οι δυνάμεις το συντομότερο δυνατόν και μάλιστα με ε, στρατιωτική ε, και μη στρατιωτική συμμετοχή. Είναι πολύ σημαντική η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοινωνικών χωρών της ε, στο πλαίσιο της ε, στρατιωτικής ανάπτυξης. Ε, το κλίμα και οι φυσικές καταστροφές θα δημιουργήσει ενδεχομένως προσωρινή αλλά και μόνιμη μετανάστευση και πρέπει να προσαρμοστούν οι πολιτικές στα σύνορα ώστε να υπάρχει η κατάλληλη ετοιμότητα σε περίπτωση ανθρωπιστικής κρίσης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Νικολάη. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να κάνω πολιτική δήλωση, γιατί η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να είναι πολιτική η προσέγγιση της έκθεσης αυτής. Συμφωνώ με την προσέγγιση της, της προσέγγισή σας σε γενικές γραμμές. Θεωρούμε ότι είναι μια καλή αφετηρία για τη συζήτηση και για ανταλλαγή απόψεων. Εμείς θα υποβάλουμε και τροπολογίε, αλλά θα ήθελα να σας ζητήσω να είστε λίγο πιο ρεαλιστείς. Είναι δύσκολο η κρίση να μετατραπεί σε ευκαιρία σε αυτή την περίπτωση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο επίσης να θέσουμε και προτεραιότητες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Ένα ερώτημα θέλω να σας θέσω αυτό που είπατε για τη θεσμική δημιουργικότητα και την ανάγκη θεσμικής δημιουργικότητας. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να αναπτυχθούν ε, οι υπάρχουσες υποδομές, ε, όμως πρέπει να λειτουργεί καταρχάς αυτή, να λειτουργούν καταρχάς αυτές οι υποδομές. Τι εννοείται European Engineer Corps? Τι εννοείται όταν προτείνεται ένα τέτοιου είδους ε, σώμα. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ. Εγώ καταρχάς να ευχαριστήσω και να συμφωνήσω με την εισηγήτρια που είπε ότι πρέπει να είμαστε πολύ ρεολοι πραγματιστές. Η συνάδελφος Νικολά είπε ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Πραγματικά πρέπει αυτό να διέπει όλη την έκθεση και να το θυμόμαστε αυτό πάντοτε. Έχουμε την ε, Επίτροπο Γεωργίευα, η οποία ε, ε, ήδη στο τσουνάμι το 2004 διασφάλισε να έχουμε ενεργό δράση. Επίσης, ανθρωπιστική δράση στη Λιβύη είχαμε γενικά Νομίζω ότι έχουμε μια συνολική προσέγγιση σε στρατιωτική και μη στρατιωτική βάση. Κάθε φορά που έχουμε αυτές τις κρίσεις και φυσικές καταστροφές και είτε πρόκειται για μια φυσική καταστροφή ή ε, ανθρωπογενή καταστροφή, ε, μπορούμε να βοηθήσουμε ανεξαρτήτως του ε, παράγοντα που προκαλεί την καταστροφή. Επίσης, ε, στο σημείο 14 έχουμε ένα κατάλογο ε, περιοχών και χωρών που είναι πιο ευάλωτες στην αλλαγή του επόμενες δεκαετίες. Αυτό υπάρχει ήδη. Πρέπει λοιπόν να δούμε γενικά τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει, να κοιτάξουμε πού υπάρχουν προβλήματα. Στο 15 ένα έγγραφο πολιτικής ε, για μια ε, ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας του κλίματος. Νομίζω ότι έχουμε ε, εργαλεία με τα οποία μπορούμε να αντιδράσουμε όταν υπάρχει μια ανθρωπογενής ή φυσική καταστροφή. Όμως, το να τα ονομάζουμε όλα αυτά ως μια ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας του κλίματος, έτσι με τόσο ε, δεν ξέρω, στυλιζαρισμένο τρόπο. Ε, είναι ένα έγγραφο και πολύ απλό και θα ήθελα να μην έχουμε τόσο μεγαλόστομες δηλώσεις, ε, να μιλάμε για ρεαλισμό και πραγματισμό. Ναι, ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα σήμερα, ξέρουμε, τα κατονομάζουμε και θα αντιδράσουμε καταλήλως. Αλλά τώρα να χρησιμοποιούμε τέτοιες πομπόδεις εκφράσεις δεν το συμβουλεύω. Και αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία θα έπρεπε να πάει και η έκθεση, αλλά και οι τροπολογίες να συνάδουν με την πραγματικότητα. Bien, Αν δεν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο, κύριος Τάραντ, ε, για ένα πρώτο συμπέρασμα. Πάρα πολύ προσεκτικός θα είμαι εγώ στην εξαγωγή συμπερασμάτων σε αυτή τη φάση. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα σχόλια και την κριτική τους. Εγώ θα ήθελα να προσπαθήσω να απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας Νικολάη με το θέμα του European Engineer Corps. Θα το χρειαστούμε στο μέλλον. Αλλά εγώ δεν είμαι βαθμός για να μπορώ να σας εξηγήσω πώς ε, θα λειτουργεί αυτό το πράγμα. Και εγώ θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες. Σαν μια επιτόπου τέλος πάντων υποδομή, ή ένα αεροδρόμιο. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, να συζητάμε για το θέμα της ε, κλιματικής αλλαγής ε, και να βάζουμε πάρα πολλά πράγματα συζητώντας αυτό το θέμα. Και συμφωνώ θα μπορούσε να είναι να περιλαμβάνει λιγότερη πολιτική ιδεολογία το, ε, η έκθεση, όπως είπε και η συνάδελφος από το ΕΛΚ, αλλά δεν ξέρω την πολιτική ή την ιδεολογική πλευρά να μειώσω. Τέλος πάντων θα λάβω υπόψη το σχόλιο σας παρόλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Θα περιμένω εν αγωνίω στην περαιτέρω συνεργασία μου με τους κοιόδης εισηγητές. Bien. Euh, et donc nous avons euh, des amendements qui peuvent être déposés jusqu'au 4 euh, euh, Μέχρι τις 4 Ιουλίου προθεσμία υποβολής τροπολογιών, οπότε σας καλώ να συνεχίσετε τη συζητήσή σας, γιατί αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να περάσουμε τώρα στο τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξής μας, που είναι μία ακόμη έκθεση του κυρίου Πάσκου. Για τις ρήτρες αμοιβαίας άμυνας και αλληλεγγύης που έχουν συμπεριληφθεί στη συνθήκη της Λισαβόνας. Πολιτική και επιχειρησιακή διάσταση. Είναι γεγονός ότι δεν είναι μόνο θεωρητική η συζήτηση. Θα θέλαμε να είναι μόνο θεωρητική. Αλλά είναι και θέμα δόγματος, το οποίο κατά κάποιο τρόπο παραγνωρίστηκε κατά τη σύνταξη της ε, συνθήκης της Λισαβόνας ε, δεν είναι επανάσταση, αλλά είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη ε, στην ε, πολιτική ε, κοινή άμυνα. Και αν στα κράτη-μέλη υπήρξαν πάρα πολλά εργαστήριο για τις μόνιμες συνεργασίες στο πλαίσιο της συνθήκης, της Λισαβόνας, αυτό το θέμα δεν έχει εξεταστεί ει βάθος ακόμη και ελπίζουμε ότι αυτή η έκθεση θα δώσει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί από αυτού του πολύ σημαντικού ζητήματος. Κύριε Πάσκου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι κάτι το οποίο άρχισε με ένα ερώτημα. Αν κάποιο κράτος μέλος ζητούσε την εφαρμογή των άρθρων αυτών, τι θα γινόταν. Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα το οποίο θέσαμε και προσπαθήσαμε να απαντήσουμε. Όμως, Εμείς τελικά τι κάναμε, προετοιμάσαμε ένα έγγραφο εργασίας και το μοιράσαμε στους σκιώδεις εισηγητές και κατόπιν συζητήσεων με, με ε, συναδέλφους, ε, με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου που έχουν ευθύνες ε, σε περίπτωση ενεργοποίησης τέτοια ρήτρα. Πρέπει να φτάσουμε σε ένα πρώτο σχέδιο εγγράφου, το οποίο θα το διανύμω στους συναδέλφους. Στις 31 Ιουλίου πρέπει να έχουμε τις μεταφράσεις έτοιμες. Μετά ξέρετε ότι η εξέταση του ε, σχεδίου της έκθεσης θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου και η προθεσμία υποβολής τροπολογιών θα είναι 20 Σεπτεμβρίου. Μετά συζήτηση της έκθεσης ε, ουσιαστικά θα την έχουμε πια τον Νοέμβριο. Τέλος πάντων αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε. Προσπαθούμε καταρχάς να αξιολογήσουμε το πλαίσιο. Γιατί αυτές τις δύο ρήτρε πρέπει να τις τοποθετήσουμε σε ένα πλαίσιο. Και το πλαίσιο αυτό δείχνει νέες απειλές και νέους κινδύνους που ενδεχομένως μπορεί να υπερβούν τις δυνατότητες μιας μεμονωμένης χώρας αν δεν υπάρξουν οι απαραίτητες διαδικασίες και τα απαραίτητα μέσα για να μπορέσουμε να ε, ε, να εφαρμόσουμε όντως στην πράξη τις ρήτρες, τότε θα είναι απλώς, συμφωνή, θα είναι απλώς ε, ε, συμβολικό. Από τη συνθήκη των Βρυξελών το έχουμε κληρονομήσει αυτό το πράγμα, όλο το σέρναμε από τότε και Το παραπέμπαμε στο ΝΑΤΟ για τις χώρες που συμμετέχουν και στους δύο οργανισμούς, όμως υπάρχουν χώρες που δεν είναι μέλη και στους δύο οργανισμούς. Και τότε δεν θα υπάρχει συμφωνία στο ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εμπλακεί αν οι χώρες ζητήσουν μια τέτοιου είδους ενεργοποίηση. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι ρήτρε ε, πηγαίνουν μαζί, για λόγους ανάλυσης τις διαχωρίσαμε και προσπαθήσαμε να έχουμε μια αντιπαράθεση. Από τη μία είναι το πεδίο εφαρμογής, από την άλλη είναι οι δυνατότητες και από την άλλη είναι οι δομές και οι διαδικασίες. Αφού αξιολογήσουμε το ρόλο των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, υπάρχει αυτή η ιδέα αυτού που προτείνεται και στη δική σας έκθεση, να έχουμε ένα μόνιμο ε, αρχηγείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο. Πρέπει να δούμε πώς, μπορεί να, πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε κάποιες αντιδράσεις που υπάρχουν από κάποιες χώρες. Σε ό,τι αφορά τη ρήτρα αλληλεγγύης. Δεν ακούσαμε το αστείο από τον κύριο Γκάλερ. Δυστυχώ δεν ακούσαμε την αρχική, το αρχικό αστείο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη ρήτρα αλληλεγγύη. Σίγουρα υπάρχει η θέληση από τις ε, χώρες να βοηθήσουν να συνδράμουν την πτυτόμενη χώρα. Αυτό μπορεί να δρομολογηθεί, αυτή η προσπάθεια μπορεί να δρομολογηθεί τη στιγμή που η καταστροφή ε, ξεπερνάει κατά πολύ τι ικανότητε μιας χώρας να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της καταστροφής αυτής. Και θα πρέπει να έχει αρκετή ευελιξία, ούτω ώστε να λάβει υπόψη διάφορες περιπτώσεις για να είναι αποτελεσματική και να βοηθάει πραγματικά τις ε, χυμαζόμενε χώρες. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι οι χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν τα κενά τους. Πού τους λείπουν τα μέσα ε, γιατί αλλιώς ε, θα υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί ε, θα ξέρουν α πούμε ότι εκεί που έχουν κενά αυτοί κάποια θα τα καλύψουν μονίμως ε, λόγω της ρήτρα αλληλεγγύη και δεν πρέπει να είναι σωστό αυτό, δηλαδή τα, καμία, κάποια χώρα να μην κάνει τίποτα. Επομένω, αυτή η προσπάθεια ανταπόκρισης με ή χωρίς την προσφυγή στην ρήτρα πρέπει να δούμε ποια είναι η εσωτερική στρατηγική ασφάλεια, πρέπει να αξιολογήσουμε την, ε, το δυναμικό τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση. πρέπει να τα αξιολογήσουμε όλα αυτά. Και το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τον κατακαιρματισμό, γιατί υπάρχει κατακαιρματισμό. Θα πρέπει να αποφύγουμε τι περιττέ επικαλύψει και θα πρέπει να εξορθολογήσουμε και να πλουστεύσουμε τι διαδικασίε που είναι τεράστια σημασία. Υπάρχουν δύο ε, απόψεις. Η μία λέει ότι θα πρέπει όλα να τα βάλουμε σε ένα τίτλο, να είναι μία ας πούμε ενότητα, μία θηρίδα και άλλες απόψεις, η άλλη άποψη λέει ότι πρέπει να υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ των μεν και των δε. και ανάλογα με την φύση της κατάστασης να δώσουμε προτεραιότητα στον ένα ή στον άλλο τομέα. Δηλαδή άλλο είναι η φυσική καταστροφή και άλλο είναι η μετανάστευση και το πρόβλημα λόγω μετανάστευση. Πάντως, όταν μιλάμε με τους εμπλεκόμενους αυτέ αυτές τις καθημερινά, μαθαίνουμε ότι καμία κρίση δεν είναι μονοδιάστατη. Όλες οι κρίσεις έχουν διάφορες διαστάσεις. Επομένως, χρειάζεται κάποιο συντονισμό πάντα. Ένα άλλο στοιχείο είναι πώς θα βελτιώσουμε τον πολιτικό συντονισμό ε, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Γιατί είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να έχουν στενή επαφή και εδώ ξέρετε ότι ο μηχανισμός θα πρέπει να λειτουργεί ομαλά. Η πρόθεσή μας και αυτό που είπαμε στους κοιόδης συζητητές είναι να υπάρχει ενημέρωση σε κάθε φάση της διαδικασίας. Θα ενημερώνουμε τους σκιώδεις σε κάθε φάση από εδώ και πέρα και τους ανθρώπους με τους οποίους ήρθαμε ε, σε επαφή για να γράψουμε την έκθεση. Αποκλείεται να θεωρηθεί αυτό, αυτή η έκθεση, αυτό το κείμενο ε, μυστικό ε, και να το παρουσιάσουμε έτσι ευνίδια. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Θέλουμε να βρούμε κάτι το οποίο θα είναι και λειτουργικό και θα ικανοποιεί όλους μας. Ευχαριστώ για τις πρώτες αυτές απόψεις που μας είπατε. Είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε. Θα θα κάνουμε τα πράγματα με άνεση χρόνου. Ε, οι προθεσμίες είναι καλές. Είναι μια προκαταρτική ε, αυτή η συζήτηση. Κυρία Γιαννάκου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και τον εισηγητή με τον οποίο είχαμε ε, μια πρώτη συνάντηση σκιώδης συζητητές. Ε, η ρήτρα αυτή αλληλεγγύης και στο επίπεδο της άμυνας και στο επίπεδο ε, της, αλληλεγ... της ε, περίπτωσης τρομοκρατικών επιθέσεων ή και άλλων ε, παραδείγματος χάρη φυσικών καταστροφών κτλ είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να σας πω ότι το επεξεργαστήκαμε στην συνέλευση και δεν είναι εδώ ο κύριος Μπρόκ αλλά η πρόταση αυτή ήταν δική μου πρόταση την οποία συνυπέγραψε και ο κύριος Μπρόκ, την κάναμε μαζί και νομίζουμε ότι έχει τεράστια σημασία διότι μπορεί αφενός να βοηθήσει ε, στη λογική ε, της δημιουργίας των προϋποθέσεων <coughs> για ένα ευρωπαϊκό αμυντικό σύστημα ενώ ταυτόχρονα όπως και ο κύριος Πασκού στην ε, έκθεσή του αναφέρει ε, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχώρηση του ΝΑΤΟ από τους σκοπούς και τις διαδικασίες για τις οποίες έχει ταχθεί. Και αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα υπάρχουν δύο πλευρές του ζητήματος βέβαια υπάρχει το άρθρο 42.7 της συνθήκης που αναφέρεται στην περίπτωση που υπάρχει κάποια επίθεση στο έδαφος μιας χώρας. Και υπάρχει και η ρήτρα αλληλεγγύης ε, η οποία αφορά στο άρθρο 222. Ε, το ερώτημα πάντοτε είναι αν διάκριση θα γίνει ανάλογα με τη χώρα η οποία μπορεί να επιτεθεί θεωρητικός η Ευρώπη δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται επίθεση όπως έχουν τα πράγματα σήμερα σε διπλωματικό επίπεδο. Αλλά οι προβλέψεις πάντοτε πρέπει να υπάρχουν ε, στα θεσμικά κείμενα. Ε, και επομένως ε, αυτό που πρέπει να είναι σαφές είναι πως πρέπει και η ρήτρα για την άμυνα και η ρήτρα αλληλεγγύης να είναι πάντοτε ανεξάρτητες από το ποιος ε, κάνει την επίθεση ή τι είδους επίθεση είναι. Επομένως πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό κάπως πιο αυτοματοποιημένο για να μπορεί να παίρνει ε, τις ανάλογες αποφάσεις γιατί είναι βασικά πολιτικό ζήτημα. Ε, εδώ υπάρχει ένα ερώτημα πώς θα διαμορφωθεί κατά κάποιο τρόπο η επιχειρησιακή ηγεσία ή το όποιο σύστημα θα εισηγείται για την απόφαση. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε αυτό είναι βέβαια και θέμα του ε, ΣΟΜΕ, του, της Συνόδου Κορυφής. Ε, θα είναι παραδείγματο χάρη το Συμβούλιο κατευθείαν, ε, θα είναι η Υπουργοί Εσωτερικών, θα είναι η Επιτροπή ε, η πολιτική και η Επιτροπή Ασφάλειας και αυτό πρέπει να εξεταστεί. Συμφωνώ επίσης με τον εισηγητή ότι ε, ενώ δεν υπάρχει κάποιο κείμενο αναφοράς αυτή τη στιγμή, είναι δηλαδή αρχίζουμε εμείς πρώτοι, ε, αυτά πρέπει να γίνουν με διαφάνεια, με πλήρη διαφάνεια. Είναι κάτι σημαντικό που μπορεί αυτή τη στιγμή ε, να φαίνεται απίθανο ή αχρίαστο αλλά μπορεί να αποτελέσει ένα καλό εργαλείο που θα βοηθήσει στην αλληλεγγύη των κρατών μελών, θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να ασκήσουν κοινέ πολιτικές και μπορεί να βοηθήσει και σε αυτό που μακροπρόθεσμα πάντοτε είχαμε θέσει, δηλαδή ε, τη δημιουργία τέτοιων μηχανισμών ακόμη και στην ε, παραγωγή των οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν πάρα πολλά κεφάλαια ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως έχει πολλαπλό ενδιαφέρον και βεβαίως συνδέεται ε, και με την λειτουργία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης αλλά ουσιαστικά μπορεί και πρέπει να συνδεθεί ε, με όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια των χωρών των κρατών μελών και με τις οποιασδήποτε εξωτερικές απειλές ε, αυτές που γνωρίζουμε και πιθανόν και αυτές που δεν έχουμε γνωρίσει ακόμα. Γιατί παραδείγματο χάρη αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό ο κύριος εισηγητής, κάποτε αυτό δεν αποτελούσε πρόβλημα. Σήμερα ε, δημιουργούνται διάφορα ζητήματα για την Ευρώπη και πρέπει μέσα στα πλαίσια των δημοκρατικών θεσμών και των αρχών και αξιών βέβαια στις οποίες βασίζεται ε, η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα βασίζεται πιστεύω και η εξέλιξή της ε, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τους μηχανισμούς εκείνους που θα εξυπηρετούν ε, θα εκφράζουν την αλληλεγγύη των κρατών μελών άρα και των λαών θα εκφράζουν την ανάγκη των πολιτών για ασφάλεια, γιατί αυτή γίνεται όλο και ισχυρότερη, η ανάγκη των πολιτών, και βέβαια θα συνδέουν τα συστήματα έτσι, ούτω ώστε σιγά σιγά να δημιουργηθούν και άλλες προϋποθέσεις που εξαιρετικά μας ενδιαφέρουν από πλευράς κοινής δράσης. Χωρίς, όπως είπα, όπως αναφέρει και ο εισηγητής, ε, να απομειώνεται ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην περίπτωση αυτή. Επομένω, θέλω να συγχαρώ για το κείμενο τον εισηγητή και νομίζω ότι έχουμε όλο το χρόνο να προχωρήσουμε ε, μαζί, να συζητήσουμε αρκετά εδώ ε, και να συνεννοηθούμε. Είναι μια πρωτοβουλία στην ουσία που έχει τεράστια σημασία για το Κοινοβούλιο διότι υπάρχουν και τα ζητήματα του πώς ελέγχονται όλα αυτά από πλευράς Κοινοβουλίου και νομίζω ότι μετά το Σεπτέμβριο και αφού παρουσιαστεί όπως είπε ο εισηγητής τον Ιούλιο το πρώτο, η πρώτη πρόταση ε, θα μπορέσουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο, με συνεννόηση να προχωρήσουμε στην απόφαση για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Merci. Ε, Ευχαριστώ. Ε, Καλημέρα. Συμφωνώ ότι είναι πολύ σημαντική η έκθεση αυτή και ανησυχώ ότι θα δούμε μόλις στα τέλη του Ιουλίου το σχέδιο όπου οι σημαντικοί άνθρωποι θα είναι διακοπές. Πάντως είναι μια έκθεση που πρέπει να διαδοθεί όσο γίνεται περισσότερο στο Κοινοβούλιο. Να, την, να φτάσει σε πολλούς και επίσης και στην Κομισιόν και σε στενή συνεργασία με την Κομισιόν να την συντάξουμε και βέβαια και με το ΝΑΤΟ. Να φτάσει και στο ΝΑΤΟ, γιατί το ΝΑΤΟ γνωρίζει πολλά για το δυναμικό των ευρωπαϊκών κρατών να αντιδράσουν σε όλα τα ενδεχόμενα. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να αξιοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες που έχει το ΝΑΤΟ και την εμπειρία. Όσο μπορούμε. Ένα διαδικαστικό ερώτημα, Πρόεδρε. Η Επιτροπή ΑΦΚΟ, συνταγματικών υποθέσεων δηλαδή, σκεφτόταν να ετοιμάσει μια γνωμοδότηση για αυτό το θέμα. Καλή ιδέα μου φαίνεται. Και εγώ στην ΑΦΚΟ υποστήριζα ότι πρέπει να κάνει μια τέτοια η Επιτροπή Συνταγματικών ε, Υποθέσεων για να εξετάσει τις θεσμικές πτυχές από την εφαρμογή αυτών των ε, ρητρών. Ίσως να μην υπάρχουν. Πάντως είναι ένα θέμα που καλό θα ήταν να διαρευνήσουν στην ΑΦΚΟ. Επίσης, στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, Ξέρουμε στικτοδός ότι δεν υπάρχει μία λύση κατάλληλη για όλα τα κράτη-μέλη, μία λύση για όλα τα ενδεχόμενα, για όλες τις περιπτώσεις. Το είπε και ο εισηγητής. Και καθώς εξετάζουμε το άρθρο 222 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 4270, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τρία είδη ενισχυμένης συνεργασίας ε, με βάση τη συνθήκη στην ΚΠΑ, όπου ομάδες κρατών μπορούν να προχωρήσουν περισσότερο και γρηγορότερα από τους υπόλοιπους, από τη βάση ας πούμε. Και υπάρχει και η τακτική ενισχυμένη συνεργασία υπό το 3.29, παράγραφος 2 και το άρθρο 44 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που μιλάει για τα ειδικά καθήκοντα και τις ειδικές αποστολές που μπορεί να προωθήσουν μία ομάδα κρατών και το άρθρο 46 που είναι η μόνιμη συνεργασία, οι μόνιμες δομές συνεργασίας. Το άρθρο 329 είναι από τη Συνθήκη Λειτουργίας Ευρωπαϊκής. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε σε αυτή την έκθεση τη δυνατότητα και πιθανότητα να υπάρχουν τέτοιες ομάδες κρατών που θα δρούν και ομάδες κρατών που θα άδρανουν, που δεν θα συμμετέχουν σε όλες τις περιπτώσεις. Τώρα για το έγγραφο που μας ετοίμασε ο κύριος Πάσκου και τα όσα μας είπε στην παρουσίασή του. Δεν συμφωνώ τη συμπερίληψη των δύο αυτών ρητρών στη συνθήκη της Λισαβόνας. Ήταν απλώς μια συμβολική χειρονομία. Αν θυμάμαι καλά, δεν επετέφερε αυτό έτσι εύκολα και ανέξοδα. Η συνέλευση δεν συμφώνησε τόσο εύκολα να συμπεριληφθούν αυτές οι ρήτρες για να κλείσει έτσι η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, παρότι δεν το περιμέναμε, αποδείχτηκε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το διαπραγματευτούμε αυτό το σημείο. Είναι λάθος λοιπόν το Κοινοβούλιο να είναι τόσο κομπορήμων για τη συμπερίληψη αυτών των δύο ρητρών. Αντίθετα, είναι μια ε, ουσιαστική και ποιοτική βελτίωση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και του δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιτρά στο, στις πολιτικές ασφάλειας και άμυνας. Και αν λειτουργήσουν, ε, η ολοκλήρωση του τομέα της ασφάλειας και άμυνας θα γίνει κινητήρια δύναμη για την Ευρωπαϊκή Ενότητα. Μια ένα, μια κινητήρια δύναμη που δεν έχουμε ίσως σε άλλους τομείς της πολιτικής μας. Στην στο νομικό τομέα, ας Ο κύριος Πάσκου μπορεί να μου πει τι πιστεύει ότι η Κομισιόν και η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος σκοπεύουν να κάνουν ούτως ώστε να έχουν έναν ε, εφαρμοστικό και εκτελεστικό μηχανισμό για τη ρήτρα αλληλεγγύης. Γιατί ό,τι και να κάνουμε εμείς πρέπει να δουλεύουμε προς την κατεύθυνση της Κομισιόν. Και επομένως θα πρέπει να συντονίσουμε την προσέγγιση μας με την Κομισιόν. Επιπλέον, μιλάτε για την ανάγκη πολιτικού συντονισμού σε υψηλό επίπεδο, αν θέλουμε να πετύχουμε οτιδήποτε σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα. Μπορεί να, έχει, να είναι δύο ειδών όμω. Μπορεί να είναι διαχείριση, γρήγορη διαχείριση των κρίσεων ή μια μόνιμη πολιτική δέσμευση σε υψηλότατο επίπεδο. Δεν είναι κατά ανάγκη το ίδιο πράγμα. Και δεν ε, χρειάζεται πάντα η ίδια ανταπόκριση, η ίδια απάντηση. Θεσμική, στρατιωτική. Τελευταίο μου σημείο. Λέτε πολύ σωστά ότι το ΝΑΤΟ, στο ΝΑΤΟ μπορεί να υπάρχουν καταστάσεις όπου δεν υπάρχει συμφωνία για μια συλλογική δράση. δεν συμφωνούν στον ΝΑΤΟ, ας πούμε. Αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι να συμφωνήσει το ΝΑΤΟ ότι δεν θα εμπλακεί κάπου. Επομένως, το σημείο αφετηρίας δεν είναι η διαφωνία στο ΝΑΤΟ, αλλά μέσω μιας επικοδομητικής συμφωνίας, ότι δεν θα αναπτύξει τις δυνάμει του τον ΝΑΤΟ. Δεν θα κάνει τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι παρούσα στις διαπραγματεύσεις νατοικές. Γιατί θα είναι ο προπομπός, η προπαρασκευαστική δουλειά για κάτι που θα πρέπει εν συνεχεία να ολοκληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα χρειάζεται στενή συνεργασία μεταξύ ημών και του ΝΑΤΟ. Κάπως θα πρέπει να προκύψει αυτή η συνεργασία. Πρέπει να υπάρχει ένας επιχειρησιακός μηχανισμός που θα μας βρίσκει σύμφωνους και μας και που θα αφορά αυτές τις δύο Υπόσχομαι να, σας, να σας επαφή μαζί σας και κάτι τη διάρκεια των θερινών διακοπών ε, για το σχέδιο του κειμένου. Ευχαριστώ κύριος Γκάλερ. <coughs> Ευχαριστώ. Να κάνω μια σύντομη πολιτική παρατήρηση. Θεωρώ ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να δεχτούμε πολιτικά και πρέπει να επικεντρωθούμε στο ακόλουθο όλοι οι ευρωπαϊκοί ε, πολίτες να έχουν, ευρωπαίοι πολίτες να έχουν την ίδια ισότιμη ασφάλεια. Και αυτό πρέπει να το εκφράζουμε ξεκάθαρα και να πούμε και πώς μπορούμε να το πετύχουμε καλύτερα. Ας πούμε, στις Βρυξέλλες, στο Ταλίν, στο Λονδίνο, στο Βουκαρέ, Βουκουρέστι, στο Βερολίνο, όλοι πρέπει να έχουν την ίδια ασφάλεια από άποψη Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως κάποιος ας πούμε στη Φιλανδία, στη Μάλτα ή όπως κάποιος ε, και στην ε, Λευκοσία. Ε, στη Λεμεσό. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε πολιτικά στο μυαλό μας και με αυτόν τον τρόπο να εκτελούμε το καθήκον μας. Επίσης κάτι άλλο που πρέπει να σκεφτούμε είναι κάτι που ε, πολλές φορές συζητείται στο ΝΑΤΟ και μετά απαντάνε με όχι. Το θέμα μιας ε, ε, επίθεσης στον κυβερνοχώρο είναι θέμα του άρθρου 5 στο ΝΑΤΟ. Πολλές φορές λένε όχι. Ε, ως εξέλιξη ε, αυτό το θέμα εμείς το βάζουμε σε ευρωπαϊκό πλαίσιο με το άρθρο 5 ή αντίστοιχα άρθρα. Γιατί οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ίσως θα πρέπει να γίνουν ε, αντικείμενο μιας καινούρια συζήτησης και να έχουμε και ε, κάποιες τεχνικές διαστάσεις που θα συζητηθούν ε, και να μην μένουμε σε αυτό το όχι που λέγεται συνήθως από τον ΝΑΤΟ. Ναι, δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Κύριε Πάσκου, Θέλετε κι εσείς να προσθέσετε κάτι μετά από τα όσα ακούσατε. Ε, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω στην Επιτροπή ε, γιατί καταφέραμε να βρούμε λίγη ώρα μέσα στην ημερήσια διάταξη να συζητήσουμε αυτή την προκαταρκτική έκθεση, γιατί υπάρχουν κάποια γραφειοκρατικά εμπόδια και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναφέρω. Πρέπει κάπως να πάμε παράλληλα με αυτό. Αν θέλουμε να βρίσκουμε την κατάλληλη στιγμή που η Κομισιόν θα προσπαθεί να συνθέτει Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ποια είναι η τάση στην Κομισιόν, γιατί γίνεται διαβούλευση με κάθε συμμετέχοντα και ο καθένας εκφράζει την άποψή του. Αλλά τέλος πάντων προς το τέλος του έτους οι περισσότεροι είναι πιο απεσιόδοξοι και λένε ίσως να πάμε του χρόνου. Όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάπου προς το τέλος του χρόνου, ε, ο Νοέμβριο είναι μάλλον ο, στόχος, μπορεί να έχει αρρημάσει αρκετά το θέμα και θα θέλουμε να ξανασυζητήσουμε γιατί θα θέλει το Κοινοβούλιο να έχει πληροφορίες μέσα από αυτή την έκθεση για αυτή τη διαδικασία. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι το Κοινοβούλιο θα εξετάσει αυτή την έκθεση με, σοβαρό τρόπο, σοβαρά. Κυρία Γεννάκου, συμμετέχει λίγο πολύ σε όλη αυτή τη διαδικασία, συμμετείχε στο πώς έγιναν όλα αυτά και έχει δίκιο πρέπει να δούμε ποιες ε, διαδικασίες χρειάζονται. Με ποιον ξεκινάμε. Γιατί όταν έχουμε μια τέτοια κατάσταση, ξεκινάμε με έντονα συναισθήματα, αλλά αν δεν πουλιάσουμε τα κατάλληλα κουμπιά, στο τέλος μπορεί να έχουμε ένα χάος. Όταν λοιπόν... Μάλλον συμφωνώ με τον κύριο Ντάφ και πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονό ότι κάποιε χώρε δεν θέλουν να μπουν σε αυτό. Ναι, η αλληλεγγύη είναι κάτι άλλο, αλλά όταν μιλάμε για αμοιβαία συνδρομή υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε μια κατάσταση κατά την οποία μέρος των κρατών θα αντιδράσουν θετικά. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ναι. Από την άλλη, όταν το ΝΑΤΟ λέει όχι. Η προεπιλογή είναι ότι θα μπει στο παιχνίδι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι και η κατάσταση με τις ε, συμφωνίες ε, Βερολίνο Plus. Ε, πρώτα πρέπει να πει όχι το ΝΑΤΟ και μετά είναι η ελεύθερη Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει. Και μετά ξέρετε τι γίνεται με τα μέσα και όλα αυτά. Η ίδια λογική λοιπόν πρέπει να υπάρχει και εδώ, γιατί αυτό μπορεί να συμβεί όταν έρθουμε στο προκείμενο. Η... συμβολική διάσταση δεν είναι η συμπερίληψη στην ε, συνδίκη της Λισαβόνας. Χωρίς τις απαραίτητες επιχειρησιακές δυνατότητες, ο μηχανισμός συνεργασίας θα παραμείνει μια παρέστηση, ένα όραμα ανεκπλήρωτο. Σχετικά με τα σχόλια του κυρίου Γκάλερ. Θυμάμαι ότι υπήρξε μια συζήτηση για τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, το άρθρο 5 και το άρθρο 5. Η ιδέα του να γράψω κάτι στην άκρη για αυτό το άρθρο 5, η, το συμπέρασμα ήταν ότι το άρθρο 5 έπρεπε να μείνει ως έχει, γιατί σε πολλές περιπτώσεις το ΝΑΚ θα έχει την ερμηνεία. Αν βάζουμε... Αν αρχίσουμε να βάζουμε μπαρόκ πράγματα σε αυτό, τότε ότι δηλαδή τα ιδρυτικά μέλη είναι αυτά που θα ε, εφαρμόζουν, ε, τότε φεύγουμε από τη συνθήκη και δεν έχει και εφαρμογή. Όπως και να έχει, ε, πρέπει να κάνουμε την ερμηνεία και να μείνει το άρθρο 5 ως έχει. Μία ένοπλη επίθεση ε, δημιουργεί καταστροφή. Μία επίθεση στον κυβερνοχώρο απλώς διακόπτει τον ε, ε, φυσιολογικό ρουν των γεγονότων. Έτσι λοιπόν είναι σαν μια κουφιά βόμβα, πώς να το πω. Από νομική άποψη λοιπόν γίνεται μεγάλη συζήτηση αν ε, κάτι εφαρμόζεται όχι από αυτή την άποψη. Αλλά τέλος πάντων θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω για τη συμβολή σας. Ήταν μια προκαταρκτική ανταλλαγή απόψεων. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο και αφήστε με να σας πω επίσης ότι θέλουμε να δράσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται γιατί δεν θέλουμε να μην προλάβουμε την προθεσμία σε σχέση με τόσα κάνει η Κομισιόν. Θέλουμε να την παρακολουθούμε. Επίσης, όταν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, θα σας το στείλω αμέσως, αλλά και στους ε, φίλους από το Συμβούλιο και την Κομισιόν, για να μπορέσουμε να το έχουμε μπροστά μας αμέσως και να βρούμε μια λύση. Αυτά. Δεν με ενδιαφέρει τόσο αν είναι θέμα διακοπών ή όχι τότε, αν είναι περίοδος διακοπών ή όχι, είναι σημαντικό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Πριν ολοκληρώσουμε, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ε, κύριος Μουρτζόν που είναι εδώ, ήθελε να παρέμβει. Παρακαλώ. Όχι απαραίτητο. Αν είχε κάποια τεχνικά ερωτήματα το θεμα ευχαριστω πολυ ευχαριστουμε πριν ολοκληρωσουμε η υπηρεσια εξωτερικης δρασης κύριο μουρτζον που ειναι εδω ηθελε να παρεμβει παρακαλω οχι απαραιτητο αν ειχε καποια τεχνικα ερωτηματα το κοινοβουλιο για την ε, σκηνή πρόταση με την Κομισιόν, τότε θα μιλούσα. Όπως είδατε σήμερα, είμαστε σε ένα πολύ προκαταρκτικό στάδιο της συζήτησης. Ο κύριος Πάσκου και οι Σκιώδης έχουν αυτό το καθήκον να έρθουν σε επαφή μαζί σας για να συζητήσουν τέτοια θέματα. Αυτά. Ευχαριστούμε. Σας καλώ να μείνετε σε στενή επαφή για αυτό το θέμα που είναι πολύ σημαντικό και είναι πραγματικά χρήσιμο εμείς στο Κοινοβούλιο να έχουμε μια θέση επ' αυτού. Η οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει και κάποια συζήτηση στα κράτη-μέλη σχετικά με τις επιπτώσεις αυτών των ρητρών. Ευχαριστώ. 11 Ιουλίου η επόμενη συνεδρίαση το πρωί. Και έχουμε και τον ε, στρατηγό Σιρέν που θα έρθει εδώ να μιλήσει.